Επιτροπή για το θέμα της εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Επιτροπή Ισότητας των Φίλων και Δικαιωμάτων των Γυναικών. Εφιστώ την προσοχή στα μέλη ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει catch the eye ούτε και μπλε κάρτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και σαν πρώτη αγορητή θα είναι η συντάκτρια της ε, ερώτησης ε, η κυρία Γκαρθία Πέρεθ. Πέντε λεπτά έχετε τον λόγο κυρία Γκαρθία Πέρεθ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πάνω από 9 εκατομμύρια γυναικών ήταν θύματα στην Ευρώπη αυτής της βίας ε, από τους άντρες είναι δύσκολο να αναφερθούμε σε αυτόν τον αριθμό χωρίς να αισθανθούμε ντροπή. Είναι δύσκολο να πούμε αυτόν τον αριθμό χωρίς να γνωρίζουμε ότι πίσω από αυτόν τον αριθμό βρίσκονται συντετριμένες ζωές γυναίκες που δολοφονήθηκαν από το, τους σεξιστές άντρες που δολοφονούν από εκείνους που πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι αντικείμενο κυριότητάς τους επειδή πιστεύουν ότι δεν είναι λέει ε, δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των φίλων στην κοινωνία. Σήμερα 25 Νοεμβρίου έχουμε την ευθύνη μπροστά σε αυτούς τους αριθμούς και την ευθύνη να φωνάξουμε δυνατά, να αρθρώσουμε δυνατά τη φωνή μας, να αποφύγουμε τη σιωπή, τη σιγή, να δεσμευτούμε να εργαστούμε για τη μεγαλύτερη κοινωνική μάστιγα του κόσμου σήμερα, στον κόσμο και στην Ευρώπη έχουμε και πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνες μας. Είναι η στιγμή να πάψουμε τις διακηρύξεις, να σταματήσουμε λέγοντας καινούς λόγους, να αρχίσουμε να δρούμε, να δράσουμε. Δεν μπορούν να περιμένουν οι γυναίκες άλλο. Μέρα με τη μέρα βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης πώς ε, και στα τηλεοπτικά δελτία πώς οι γυναίκες συνεχίζουν να δολοφονούνται. Συντρίβονται οι ζωές τους ε, και οι ζωές των παιδιών τους, ε, αγοριών και κοριτσιών. Πρέπει να ζήσουμε σε μια κοινωνία πιο ίση, με μεγαλύτερη ισότητα. Πρέπει να υπομισθούμε τις ευθύνες μας. Είναι υποχρέωσή μας, είναι ευθύνη μας. Γι' αυτό απευθύνουμε σήμερα μια σειρά ερωτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας οδηγεί αυτό το θέμα στη συζήτηση επ' αυτού στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναμένουμε να υπάρξουν δεσμεύσει και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσει για το έργο που πρέπει να επιτελεστεί στο μέλλον. Να γνωρίζουμε πότε θα υποβάλει την πρόταση για τη στρατηγική της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη τοποθετηθεί επί του θέματος πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η στρατηγική. Για μας είναι θεμελιώδους σημασίας ότι μεγάλο μέρος της στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει πρέπει να αποτελεί η καταπολέμηση της βίας του φύλου εις βάρος των γυναικών αλλά και άλλα πράγματα. Έχουν γίνει βήματα από τα θεσμικά όργανα σε αυτό το θέμα. Η εντολή προστασίας των θυμάτων ήταν θεμελιώδες στοιχείο Λιγότερο από ένα χρόνο πριν <clears throat> υλοποιήθηκε, ε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την μετάθεση στο νομοθετικό πλαίσιο αυτών των προτάσεων. Πότε θα μας υποβάλει την αξιολόγησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς λειτουργήσε αυτή η εντολή προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα νομοθετικά, υποχρεωτικά και οπωσδήποτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που διεκδικούμε αυτό το θέμα από το Ευρωκοινοβούλιο. Όχι μόνο με μέτρα υποστήριξης από οργανώσεις και προγράμματα για τις γυναίκες. Δεν θα επιλύσουμε τα προβλήματα μόνο με αυτόν τον τρόπο. Είναι αναγκαίο να νομοθετήσουμε. Διότι η νομοθεσία είναι δέσμευση. Είναι η νομοθεσία μια υποχρεωτική εφαρμογή της νομοθεσίας και των μέτρων από τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών. Ακούσαμε πολλές φορές να μας λένε ότι δεν υπάρχει λέει, επίπεδο αρμοδιότητας στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της σεξιστικής κατά των γυναικών. Δεν παραδίδουμε τα όπλα όμως, δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Αν καταφέραμε η Ευρώπη να έχει αρμοδιότητες στα θέματα της καταπολέμησης κατά της οικονομικής κρίσης, επίσης μπορούμε να αναζητήσουμε τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει η Ευρώπη για να καταπολεμηθεί η βία, η σεξιστική βία εις βάρος των γυναικών. Να είναι πιο δίκαια και ανθρωπιστική κοινωνία μας. Γι' αυτό ας αναζητήσουμε λοιπόν από το Συμβούλιο και να ζητήσουμε για την Επιτροπή Επιτροπή, εμείς ως Κοινοβούλιο να υπάρξει αυτή η νομοθετική ικανότητα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πια, δεν μπορούμε με αναγγελίες ε, και κάποιες άλλες ε, ε, αναφορές να ικανοποιηθούμε. Μιλάμε για τη ζωή γυναικών, για τη ζωή του ημίσεως του πληθυσμού της Ευρώπης. Αξίζει η, το ήμιση του πληθυσμού το σεβασμό μας. Αξίζουν οι γυναίκες το σεβασμό μας και είναι στα χέρια μας να κάνουμε πολλά περισσότερα από όσα γίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να εμπλέκει όλους και όλες. Όλα τα θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα. Είναι αναγκαίο ήδη αμέσως να ενώσουμε, να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας. Το αξίζουν οι γυναίκες αυτό. Θυμόμαστε όλες εκείνες που δολοφονήθηκαν από τους ε, τρομοκράτες, ε, ματσιστές, ε, σεξιστές άνδρες και κάνουμε λόγο για το μέλλον της δικής μας γενεάς αλλά και των κορών μας, των θυγατέρων μας. Είναι υποχρέωσή μας αυτό και πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Σα ισπανικά σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Επιτροπής η κυρία Γιούροβα παρακαλώ έχει τον λόγο. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που θέτετε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα επευκαιρία της διεθνού ημέρας για την κατάργηση της βίας κατά των γυναικών. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζουν να ενταχθούν στην ε, ημέρα ε, εκστρατείας κατάργησης της βίας κατά των γυναικών. Η βία κατά των γυναικών παραμένει πρόκληση σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το 2015 οι γυναίκες δέρνονται, ταπεινώνονται, βιάζονται, κροτηριάζονται, παρακολουθούνται, παρενοχλούνται και εξαναγκάζονται σε γάμο. Η βία συμβαίνει και μέσα στα σπίτια, από τους συντρόφους, από τα μέλη της οικογένειάς τους, στο χώρο εργασίας, στο χώρο εκπαίδευσης, από συναδέλφους, συμφοιτητές, καθηγητές ή επικεφαλής. Μπορεί να γίνει online, στους δρόμους, από ξένους. Ξέρουμε ότι μία στις τρεις γυναίκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τέτοια εμπειρία, φυσική ή σεξουαλική βία ή και τα δύο. Και η βία έχει επίπτωση καθ' τη διάρκεια της ζωής της γυναίκας στην υγεία ε, των γυναικών και στις οικογένειάς τους. Επίσης στην οικονομία και στην οικονομία συνολικά. Το να προωθήσουμε την ισότητα των φίλων και να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών είναι απαραίτητο. Οι γυναίκες θα πρέπει να ενδυναμωθούν για να φύγουν από σχέσεις όπου υπάρχει βία εναντίον τους δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται για να ολοκληρώσουν το δυναμικό τους στο χώρο εργασία και στην κοινωνία εν γέννη. Θα παρουσιάσω το Δεκέμβριο ένα λεπτομερές σχέδιο της Κομισιόν και μια δέσμευση για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων τα επόμενα χρόνια. Θα το υποβάλω και στην Επιτροπή Γυναικών. Αυτή τη στρατηγική δηλαδή για την ισότητα των φύλων για τα έτη 2016 μέχρι 2019. Συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς και μαζί σας και η συνεισφορά σας ήταν πολύτιμη. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι περαιτέρω μέτρα για να υποστηρίξουμε τα κρατη για να καταπολεμήσουν και να προλάβουν ε, όλες τις μορφές βίας λογοφύλου. Η, αυτού του τύπου η βία ε, αντιμετωπίζεται από την Κομισιόν με μια ευρεία προσέγγιση που θα βασίζεται στην νομοθεσία, στην αφύπνιση, στη βελτίωση της γνώσης και της, συλλογής των δεδομένων. Θα εστιάσω καταρχάς όμως στην νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε νομοθεσία για να παρεμποδίσει τη βία κατά των γυναικών και να προστατεύσει και να υποστηρίξει τα θύματα καθώς και σε περιοχές σε τόμεις όπως σε σεξουαλική παρενόχληση, ε, εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση, παιδιών και παιδική πορνογραφία. Τα δικαιώματα των θυμάτων ε, με βάση την ε, οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων ε, εξασφαλίζονται χάρη στη θέση ισχύ της οδηγίας από τις 16 Φεβρουαρίου φέτος. Θα έχει τεράστια επίπτωση στα κράτη-μέλη, ειδικά σε αυτά όπου θα πρέπει να δημιουργήσουν ε, δομές υποστήριξης των ε, θυμάτων που είναι σημαντικότατο θέμα για να καταπολεμιστεί η βία λόγω φύλου και που δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη ακόμα. Θα πρέπει να βασιστείτε στη δική μου δέσμευση ότι η Κομισιόν θα παρακολουθεί και θα καθοδηγεί την πραγματική εφαρμογή αυτού του νομοθετήματος καθώς και του ευρύτερου νομικού πλαισίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι επαρκή μέτρα προστασίας δίδονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο και ότι εφαρμόζονται στην πράξη. Από τον Ιανουάριο του 2015 τα θύματα ε, βία στο σπίτι ε, εποφελούνται από ενισχυμένη προστασία όταν ταξιδεύουν ε, και μετακινούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολές προστασίας που εκδίδονται στην οικία χώρα μπορούν να κυκλοφορήσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενσωμάτωση και η μεταφορά είναι θεραπευτική χάρη στις διαδικασίες εφαρμογής που ξεκίνησε η Κομισιόν και έχουμε τώρα εθνικούς κανόνες που μεταφέρουν την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, που είναι μια οδηγία, και στα, σε 21 κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Επίσης, στις 9 Οκτωβρίου η Κομισιόν δημοσίευσε ένα οδικό χάρτη για τη μελλοντική προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση της Ισταμπούλ, της Κωνσταντινούπολης, της, ε, που είναι μια σύμβαση και είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και τη βία στο σπίτι. Η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση θα αντανακλά την δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διακρίσεις εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η Κομισιόν υποστηρίζει την αφύπνιση και συγκεκριμένες επιτόπιες δράσεις των κρατών μελών, της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της και των ευρωπαϊκών δικτύων. Φέτος, 8 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στην καταπολέμηση βίας κατά γυναικών υπό το πρόγραμμα ε, για τα δικαιώματα και ηθαγένειας. Επίσης, ε, καταπολεμούμε τις πρακτικές ακροτηριασμού των φύλων ε, και υποστηρίζουμε τα θύματα βίας στα πανεπιστήμια για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις ανάγκες των νεαρών θυμάτων και να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη που θέλουν να ευαισθητοποιήσουν το γενικό πληθυσμό στο πρόβλημα αυτό. Με περηφάνεια σας ενημερώνω για την απόφαση της περασμένης εβδομάδας να ε, συνταχθούμε σε νέα διεθνή, συγγνώμη, να σταματήσουν νέα διεθνή προγράμματα ε, ύψους 4,3 εκατομμύριων ευρώ ε, λόγω του ότι είχαμε προβλήματα ε, με τα δικαιώματα των γυναικών. Θα πρέπει να θέσουμε στο κέντρο το θέμα αυτό και ετοιμάζουμε μελλοντικές δραστηριότητες. Ε, καλωσορίζουμε δε τη συνεργασία σας. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λόγια για τη σημασία της βελτίωσης των γνώσεών μας για τις αιτίε της βίας λογοφύλου και να ενημερώνουμε τις γνώσεις μας. Είναι σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε την κατάσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να διατυπώσουμε και να εφαρμόσουμε καλύτερες πολιτικές. Οι υπηρεσίες μου εργάζονται με τη Eurostat και, τα, το Ευρωπαϊκό ε, Οργανισμό για την Ισότητα των Φύλων, δύο βασικούς φορείς που μπορούν να βοηθήσουν για να καλυφθούν τα κενά. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κυβερνοδία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και τις αναδυόμενες, τις νέες μορφές βίας. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις πολιτικές για τα παιδιά και την ασφάλεια των κοριτσιών από τον bullying, την κατάχρηση και την εκμετάλλευση online. Επιπλέον, η Κομισιόν ετοίμασε ε, μία έκκληση 3 εκατομμυρίων ευρώ για προτάσεις καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον γυναικών και κοριτσιών ε, που συμπεριλαμβάνει εδώ και τις νέες τεχνολογίες και εξολογούμε αυτή τη στιγμή τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε. Οι αγορητέ εξ ονόματο των ομάδων τώρα για το ΕΛΚ που θα ξεκινήσει. Η κυρία Χιμένεθ Εμπεθερή, παρακαλώ. Δύο λεπτά έχει τον λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε Γιούροβα για τη δέσμευσή σας με τα υπέρ των θυμάτων. Σήμερα είναι η μέρα κατά της βίας εις βάρος των γυναικών και ακόμα πρέπει να διερωτηθούμε γιατί αυτή η μέρα. Διότι είναι θεμελιώδες να απαντήσει και να αντιδράσει η κοινωνία. Θα πρέπει να προαθούν δράσεις αποτελεσματικές για να τερματιστεί αυτή η μάστιγα για να μην συνηθίσουμε σε αυτή την κατάσταση, στη δυναμική του δεν βλέπω, δεν ακούω και δεν λέω τίποτα. Σιωπώ. Πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σπάσει αυτό το τείχος που δημιουργείται από το φόβο σε σχέση με τα θύματα. Διότι ο θήτης αισθάνεται ισχυρός δεδομένης αυτής της κατάστασης και συνεχίζει να κακοποιεί. Και στη χειρότερη περίπτωση δολοφονεί τη γυναίκα που λέει ότι αγαπάει. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων της βίας εις των γυναικών η βία αυτή προέρχεται από τους συντρόφους των γυναικών και είναι σημαντικό τα θύματα να καταγγείλουν. Αλλά για να καταγγείλουν πρέπει να αισθανθούν ότι προστατεύονται. Γι' αυτό είμαι υπερήφανη για το ότι ξεκίνησε η εντολή προστασία των θυμάτων, ώστε να αναγνωρίζονται αυτέ ε, οι καταστάσει σε όλε τι χώρε. Προ όφελο των γυναικών και τη ασφάλειά του, που προσπαθούν να ξεφύγουν από του θήτε Πολλά πρέπει να γίνουν σε σχέση με την Ευρώπη. Γι' αυτό υποβάλλουμε αυτή την προφορική ερώτηση για να ξέρουμε ποια στρατηγική ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται μεγαλύτερη δέσμευση για να σταματήσει η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπολογίζουμε 35% των γυναικών και των κοριτσιών υφίστανται κάποιο είδου βία σωματική ή σεξουαλική κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Αυτό πρέπει να σταματήσει επιτέλου. Πιστεύω στεναρά ότι αν εργαστούμε στο πεδίο τη ε, εκπαίδευση, ε, τη παιδεία, τη προστασία των θυμάτων και καλύτερο έλεγχο κατά των θητών, μπορούμε να να αποφύγουμε αυτό τον τεράστιο πόνο που προκαλείται στις γυναίκες και στα θύματα. Η αγάπη δεν πρέπει να πονά και γι' αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και επίσης οι ανήλικοι συμπεριλαμβάνονται και χαιρετίζω αυτό το γεγονός σε νέα οδηγία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Για τρία λεπτά επόμενη αγορήτρια εξ ονόματος των Σοσιαλδημοκρατών η κυρία Αρένα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν θέλω να υπενθυμίσω τους αριθμούς. Μια γυναίκα στις τρεις σήμερα στην Ευρώπη είναι θύμα βίας. Ε, πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν ανθρώπινα όντα. Είναι οι κόρες μας, οι αδελφές μας, είναι οι γυναίκες, κύριοι, είναι οι συνάδελφοί μας, είναι άτομα που βρίσκονται γύρω μας. Μια γυναίκα στις τρεις ε, γυρνάμε γύρω μας και ε, το άτομο που είναι στα δεξιά μου, στα αριστερά μου ε, υπήρξε ή θα υπάρξει θύμα βίας. Πρέπει να μιλήσουμε για τις μορφές βίας, τις ξέρουμε τις μορφές βίας. Είναι σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές, σεξουαλικές και Έχουμε ε, τους γυναικο, γυναικοκτόνους, 7 γυναίκες ε, σήμερα πεθαίνουν με αυτόν τον τρόπο, διότι πεθαίνουν επειδή είναι γυναίκες. Ε, είναι οι ακροτηριασμοί, η γεννητική, είναι η εκμετάλλευση η σεξουαλική. Ε, φτάνει πια. Φτάνει διότι είναι ανυπόφορο να βλέπουμε σήμερα ότι στην Ευρώπη έχουμε αυτήν την χαλαρότητα σε σχέση με τις διακρίσεις. Το άρθρο 8 της συνθήκης της Λισαβόνας λέει απλώς ότι πρέπει να εγγυηθούμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Είστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεματοφύλακας αυτών των συνθήκων. Σας ζητούμε απλώς να ε, υλοποιήστε αυτές τις συνθήκες, όχι να κάνετε προγράμματα και διαβήματα, αλλά να μπορέσετε να υλοποιήσετε τις συνθήκες αυτές. Είναι πολύ πιο εύκολο να υποστηρίζει κανείς το δικαίωμα ιδιοκτησίας από το δικαίωμα στη ζωή. Σας ζητούμε να υπερασπιστείτε το δικαίωμα ζωής για όλους και για το 50% του πληθυσμού της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενα χωρίς για ένα λεπτό εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών η συνάδελφος Φων Ναι, κύριε Πρόεδρε. Από το 2004 το Κοινοβούλιο συχνά μιλάει για την βία εις βάρος των γυναικών Έχουμε προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για την άρση, την κατάρριση της βίας όλων των μορφών εις βάση των γυναικών. Έχουμε το πρόγραμμα Δάφνης στην Ευρώπη για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Τι είναι όμως βία εις βάση των γυναικών είναι κατά της βίας ιδιαίτερα εις βάρος των πιο αδύναμων, ιδιαίτερα εις βάρος των γυναικών. Φυσικά είμαστε όλοι εναντίον αυτής της κατάστασης. Αλλά για τον ΟΗΕ πολλές φορές εμείς και άνθρωποι κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Οι λέξεις κάνουν την πολιτική τελικά. Για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών επαρκεί αυτό, επαρκούν τα λόγια όχι. Αλλά να προσέξουμε Σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών, βία εις βάρος των γυναικών είναι υπάρχει βία όταν δεν μπορεί να κάνει έκτρωση μια γυναίκα διότι σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία όταν είναι θύμα βία και απαγορεύεται η έκτρωση αυτό είναι βία είναι η λάθος οδός αυτή να προστατευτούν οι γυναίκες και έτσι την βία κατά των γυναικών την απορρίπτουμε όλοι σε όλες τις μορφές για τους φιλελεύθερου, στη συνέχεια Φερχόφστατ παρακαλώ Οι συνάδελφοι ε, είναι ένα θέμα σημαντικό η βία κατά των γυναικών, η σεξιστική βία είναι επίσης ένα θέμα των ανδρών και πάνω απ' όλα είναι ε, μια επονίδιστη πραγματικότητα λυπηρή, όπως ε, είπα σε διάφορες παρεμβάσεις. Πάρα πολύ συχνά γυναίκες και κορίτσια υποφέρουν από την σεξουαλική βία, σεξιστική βία και νομίζω ότι ο σύντροφος συνήθως στις 50% των περιπτώσεων είναι ο θήτης και αυτό προκαλεί θάνατο 7 γυναικών την ημέρα στην Ευρώπη επειδή οι επιθέσεις σεξουαλικές, η ανδοοικογενειακή βία και επειδή υπάρχουν ε, ακροτηριασμοί, γεννητικοί ακροτηριασμοί. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο άνδρας έχει μια φωνή στο θέμα της βίας κατά των γυναικών. Πολύ συχνά λέμε ότι είναι απλώς ένα γυναικείο θέμα και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα ενώσο θεωρείται το θέμα αυτό γυναικείο θέμα, ανεξάρτητα από τους άνδρες. Εμείς οι άνδρες πρέπει ε, να σταματήσουμε αυτήν την βία. Η ατιμορρησία για, την, ε, για τις πράξεις αυτές βίας ε, υπήρξε στο παρελθόν για όλα τα θύματα και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών. Πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύουν τις γυναίκες, αλλά υπάρχουν πολλές άλλες που δεν έχουν τέτοια μέτρα θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Έχουμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών, να την προλάβουμε, να την αποτρέψουμε, να ε, έχουμε διώξεις κατά ε, των ενόχων, αλλά μόνο 12 κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει την σύμβαση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να κάνουμε κάτι το ειδικό, δηλαδή προσχώρηση Ευρωπαϊκή προσχώρηση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση αυτή της Κωνσταντινούπολης, ώστε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και να προστατεύσουμε πολύ περισσότερες γυναίκες και να καταδικάσουμε τις χώρες οι οποίες δεν εκπληρώνουν αυτούς τους στόχους. Μηδενική ανοχή είναι ο μόνο τρόπος. Ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα και όχι μόνο γυναίκες αλλά γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σπάσουμε τη σιωπή, να υψώσουμε τη φωνή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην αρχή της συνεδρίασης αναφέρθηκε δεν θα υπάρχουν μπλε γιατί είναι ένας γύρος για τις ομάδες μόνο. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Παρακαλούμε όλοι με δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η βία είναι μια τρομοκρατία που ασκείται σε, σε ένα καθεστώς σιγής. Το αντίτιμο είναι ανθρώπινα θύματα. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η βία εις βάρος των γυναικών. Είναι μια κατάσταση που δημιουργεί ένα πλαίσιο που υποστηρίζονται ακόμα και άνθρωποι που ε, έχουν ε, ασκήσει αυτή τη φρικτή βία και βλέπουμε ότι ο Ντομινίκ Στροσκάν και πολλοί άλλοι δημόσιοι, δημόσιοι αξιωματούχοι που ενεπλάκησαν ε, βρίσκονται σε αυτό το πλαίσιο. Ζητήσαμε να υποστηρίζονται τα θύματα και δεν θα ξεχάσουμε αυτό το αίτημα και δεν θα αμελήσουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε να προστατευτούν οι γυναίκες. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης πρέπει να επικυρωθεί. Υπάρχει εδώ το δικαίωμα να υπάρχει κατάλληλα καταρτισμένη αστυνομική δύναμη, αστυνομικοί που πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί, τα κράτη-μέλη που πρέπει να έχουν εθνικά προγράμματα για την καταπολέμηση της εξιστικής βίας και να μπορούν να εργάζονται υπεύθυνοι για τις γυναίκες πρόσφυγες όταν εκτίθενται σε τέτοιου είδους βία να μπορούν να προστατεύονται με ειδική προστασία και αυτά τα άτομα από πλευράς αυτών των δυνάμεων έχουν ειδικέ γνώσεις και μπορούν να προστατέψουν τις γυναίκες. Ακόμα και η αυτοάμυνα είναι σημαντική για αυτή την προστασία. Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας κατά της βίας που έχει επιπτώσει στη ζωή μας και να καταπολεμήσουμε αυτό το καθεστώς σιωπή που δεν ευνοεί τις καταγγελίες και να μην αφαιθεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση γιατί θα πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις βίας εις βάρος των γυναικών. Η ε, συνένεση είναι μια, ένα είδος έγκριση, η σιωπή είναι ένα είδος έγκρισης ε, σιωπηρής. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα οποία απαιτούμε. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ευχαριστώ πρόεδρο Σας ευχαριστούμε πολύ για τους πράσινους ε, για 1,5 λεπτό. Σεμπαστιά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Σήμερα το πρωί αφιερώσαμε πάνω από τρεις ώρες για μια πρωταρχική συζήτηση για τα τρομακτικά πλήγματα στο Παρίσι και τις τρομοκρατικές απειλές. Και έχουμε τώρα λιγότερο από μια ώρα για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θύματα της βίας στην Ευρώπη. Διακόπτει ο μιλητής. Μπορώ να ξαναξεκινήσω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Έλεγα, σήμερα το πρωί αφιερώσαμε πάνω από τρει ώρε σε μια πρωταρχική συζήτηση για τα θύματα των τρομοκρατικών πληγμάτων στο Παρίσι και τι απειλέ τη τρομοκρατία. Τώρα αφιερώνουμε λιγότερο από μια ώρα για τα περισσότερα θύματα τη βία στην Ευρώπη που προέρχονται από τη βία κατά των γυναικών. Που κάθε μέρα και με μεγαλύτερη ένταση, ένταση πλήττουν τα θύματα από ότι οι τρομοκρατικέ απειλέ. Να ξαναπώ του αριθμού. Μία κάθε τρει γυναίκε στην Ευρώπη έχει υποστεί αυτού του είδους βία και μία στις τέσσερις σεξουαλική βία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Ευρώπη ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα ασφάλειά μα. Πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Ακόμα κάποια κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν νομοθεσίες που αποκρύπτουν ή συγκαλύπτουν αυτή τη βία ακόμα. Με αυτή την ερώτηση που καταθέσαμε επίτροπε ζητούμε να βρεθούν λύσει, να δοθούν λύσει κατεπηγόντω, γιατί κάθε μέρα δολοφονούνται γυναίκε από κάποιου που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να τι δολοφονούν από του άνδρε που έχουν αυτή την πεποίθηση και αναγκάζονται να φύγουν, να ζητήσουν προστασία σε ένα καταφύγιο ασφαλές. Ζητάμε δράση από τις κυβερνήσει κυβερνήσεις εκείνες που δεν κάνουν το καθήκον τους και γίνονται συναυτουργοί των θητών. Υπάρχει αυτή η βία η σεξιστική. Χρειάζεται η μέγιστη προστασία από τα, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κυρία Γιούροβα, έχετε παράπονα για θέματα αρμοδιοτήτων, αλλά το είπε η συνάδελφος ε, κυρία Αρένα. Όλες οι συνθήκες της Ευρώπης λένε ότι εμείς είμαστε οι θεματοφύλοι φύλακε αυτής της ισότητας. Και ποια είναι η καλύτερη ισότητα από το να καταπολεμηθεί η βία, η βία ει των γυναικών. Πρέπει να δράσουμε, να δράσετε άμεσα. Παρακαλώ. E Σα ευχαριστώ. Στη συνέχεια για 1,5 λεπτό Αγιούτο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σήμερα η σημερινή μέρα είναι γεμάτη συμβολισμό και πρέπει να υποφεληθούμε τα κράτη να επικυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Στην Ιταλία έχουμε νόμους κατά της βίας των γυναικών και παρόλα αυτά έχουμε προβλήματα και στην εφαρμογή των νόμων και σε ό,τι εφαρμογή της ε, μιας σωστής και αναλογικής ποινή. Συχνά δεν είναι σοβαρές, αρκετά σοβαρές οι ποινές εναντίον των θητών ε, τέτοιων ε, δικημάτων. Υπάρχουν νόμοι αλλά δεν ε, εξασφαλίζουν τα θύματα. Χάρη στις προσφυγές και στη μείωση της πηγής, ποινής, τελικά οι θύτες δεν ε, εκτίουν το 100% της ποινή του και στην πραγματικότητα ε, εκτίουν ένα πολύ μικρότερο κομμάτι. Επίσης, από τη στιγμή της καταγγελία του Στόκινγκ, α πούμε, τη παρενόχληση, της παρακολούθησης, μέχρι την προσφυγή στο δικαστή, παίρνει χρόνο. Θα πρέπει να κάνουμε πρόληψη σήμερα, θα πρέπει να υπάρξει προστασία και να υπάρξει και τιμωρία. Παράλληλα, με όλα τα μέτρα, τα προληπτικά, θα πρέπει να ζητήσουμε μία ενίσχυση και αύξηση των ποινών και την βεβαιότητα ότι τελικά θα εκτείονται αυτές οι ποινές, ούτως ώστε ε, να δίδονται τελικά παραχωρήσεις στους δράστες και τελικά να επιστρέφουν σε μια ωραία και άνετη ζωή αντίθετα με τις ε, γυναίκες που είναι θύματα και που θα έχουν τα σημάδια αυτής της βίας για όλη τους τη ζωή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κυρία Γιούτο. λεπτό για την ναι, Άτκινσον, παρακαλώ. Has it occurred to this place? Ναι. Θα πρέπει καταρχάς εμείς να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη πριν δώσουμε μαθήματα σε άλλους ε, τι... για το τι πρέπει να κάνουν. Εγώ στις Βρυξέλλες, στο Στραβούργο, στο Στραβούργο και στο Κοινοβούλιο ήμουν θύμα ε, λεκτικής βίας. Ε, ως ε, ευρωβουλευτής, ε, μερικές φορές ένας άλλος ευρωβουλευτής με είπε ε, «ηλίθια βλαμμένη γυναίκα». Ε, και μέλη του προσωπικού και άλλοι συνάδελφοι, ας πούμε, μας ε, επιτίθενται ε, σωστά. Επίσης, σε μια άλλη συζήτηση πριν από λίγες εβδομάδες, ένας συνάδελφος είπε μια γυναίκα ευρωβουλευτήνα παλιογι... παλιογίνεο, ας πούμε. Είναι σωστό αυτό, είναι αποδεκτό. Επίσης, με ενόχλησε ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν πιωμένος, ε, είναι γενικά έτσι παχής και ε, πολύ σωματώδης και με παρενόχλησε εδώ ε, και στους διαδρόμους. Εάν μάλιστα, και επειδή παρέπε λιγάκι, αν έπεφτε πάνω μου θα μπορούσε να με συντρίψει. Είναι, παραδεκτά όλα αυτά. Το να μεταχειριζόμαστε έτσι, ε, έτσι τις γυναίκες φαίνεται ότι είναι αποδεκτό. Εάν εμείς ε, οι γυναίκες ε, στρεφόμαστε προς κάποιον άντρο, άντρα άνθρωπο και άντρα συνάδελφο και του λέγαμε αυτά που ακούμε εμείς, θα μας επιβάλλανε ποινές. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, τίποτα. Α, κατάλαβα πολύ καλά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τους μη εγγεγραμμένους η Νταϊάν Ντότζ παρακαλώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην σημερινή κοινωνία η βία κατά των γυναικών αποκτά μορφές όλο και πιο απαράδεκτες. Σας δούμε τις συνέπειες της εμπορίας ανθρωπίνων όντων πάνω στις ζωές χιλιάδων γυναικών που πολλούνται και τι χάνουν χρήσεων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Δέχομαι τα όσα είπε ο κ. Φερχόφστατ, ότι αυτή η βία δεν απευθύνεται μόνο στις γυναίκες, αλλά στην ημέρα αυτή της βίας κατά των γυναικών βλέπω ότι γίνεται στην Βόρεια Ιρλανδία ε, με την εισαγωγή του σχεδίου νόμου ε, για την εκμετάλλευση σεξουαλική των γυναικών και την εμπορία τους θα πρέπει να γίνει προηγούμενο για άλλα κράτη-μέλη. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να αναδείξω ε, την ε, δουλειά μιας εθελοντικής οργάνωσης στη Βόρεια Ιρλανδία που ασχολείται με το θέμα αυτό και παρέχει στέγη σε γυναίκες και παιδιά που έχουν υποστεί βία ψυχολογική, σωματική. Έτσι μπορούν ε, να συνεχίσουν την ζωή τους. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε συνάδελφε και στρεφόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι κυρία Γιούροβα, Επίτροπος, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση όλοι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε όλα τα επίπεδα πρέπει να δράσουμε. Εσείς αναφέρατε εδώ ότι η Επιτροπή είναι θεματοφύλακας των συχτικών στο, από το άρθρο 8 σχετικά με την ισότητα των φύλων. Εγώ Ανασυχώ, ασχολούμαι με την ισότητα. Θέλω να υπάρξει αποτελεσματική πραγματική ε, δράση με πραγματικά μέσα και εργαλεία. Πρόκειται να έχουμε προσχώρηση ευρωπαϊκή στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να μιλήσουμε για νέες ε, οδηγίες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Εγώ προσωπικά Δεν μπορώ να μιλήσω για τη νέα οδηγία ως κάτι που θα λύσει το πρόβλημα σύντομα. Για δείτε όλη την διαδικασία προετοιμασίας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεν την κατακρίνω, αλλά ακόμα και αν βρούμε τη νομική βάση θα χρειαστούν πολλά χρόνια ούτω ώστε να τεθεί σε ισχύ στα κράτη-μέλη ε, και να έχουμε αποτελέσματα. Ειλικρινά τώρα σας μιλάω για άλλα μέσα και δηλώνω εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την νομική βάση για την νομοθεσία διότι η βία κατά των γυναικών είναι ποινικό αδίκημα και να στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τις αρμοδιότητες που έχουν βάση του ε, ποινικού νόμου. Θα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε με την προσχώρηση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που μας δίνει τις αρμοδιότητες για να δράσουμε σε επίπεδο νομοθετικό. Αλλά αυτό που είναι πιο αποτελεσματικό μέσο είναι να επενδύσουμε τα κονδύλια, τα διαθέσιμα ε, για ε, μέτρα, για εκστρατείες, ε, για υποστήριξη των οργανώσεων της βάσης, της κοινωνίας των πολιτών, να εκπαιδεύσουμε εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες που θα βοηθήσουν περισσότερο τα θύματα της βίας και μιλώντας για άλλους πρωταγωνιστές ε, που μπορούμε να υποστηρίξουμε πρέπει να μιλήσουμε για τα κράτη-μέλη που υποστηρίζουμε αλλά ταυτόχρονα ε, τα οθούμε να ε, θέσουν σε ισχύ την νομοθεσία. Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για την κοινωνία αυτή καθεαυτή, διότι η βία κατά των γυναικών σε πάρα πολλά κράτη-μέλη ε, οδηγεί σε μια σιωπηρή αποδοχή από την κοινωνία σαν να είναι κάτι το φυσικό. Σε μερικά κράτη-μέλη, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης δέχονται σιωπηρά την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να δράσουμε προς αυτές τις κατευθύνσεις για να βοηθήσουμε και επίσης οι τοπικές κοινότητες που δεν πρέπει να είναι ε, να, τυφλές και να κοφεύουν. Ας μιλήσουμε για τα θύματα αυτά καθε αυτά κυρίες και κύριοι. Έχω τις πρόσφατες στατιστικές που μας λένε ότι μόνο 50% της βίας κατά των γυναικών δηλώνεται, δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές τα θύματα παραμένουν σιωπηλά και επειδή δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στις αρχές, δεν νομίζουν ότι οι αρχές δεν θα τους βοηθήσουν. Και η οδηγία περί θυμάτων ε, είναι αυτό το ακριβώς. Θα πρέπει να μην φοβούνται να το δηλώσουν και να περιμένουν αρκετή ε, υποστήριξη από τις αρμόδιες αρχές. Και τελευταίο σημείο, και ο κύριος Φερχόφστατ το ανέφερε, είναι οι ίδιοι οι άνδρες. Οι άνδρες οι ίδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την κατάσταση. Ήμουν στην Σουηδία πρόσφατα, έχουν πάρα πολύ καλά προγράμματα, ε, κυρίως για τους άντρες ε, που παίζουν ρόλο στην καταπολέμηση αυτής της βίας. Χωρίς την δική τους κατανόηση δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα βελτιώσουμε. Πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα που απαιτεί έναν κατάλογο πολλών μέτρων που να προέρχονται από πάρα πολλούς φορείς. Ας προχωρήσουμε ε, και δεσμεύομαι να σας μιλήσω για περισσότερες λεπτομέρειες ε, το Δεκέμβριο στην Επιτροπή ε, Γυναικών σχετικά με το τι γίνεται στην Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε. <clears throat>